Θα σας παρακαλούσα να βάλετε τα ακουστικά σας, μια και θα μιλήσω ρουμανικά. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, σου, την έναρξη τη συνεδριάσεω, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή ενίσχυση τη τρομοκρατική απειλή. Θα παρακαλέσω